και σίγουρα θα επαναξετάσουμε το θέμα και στην Κομισιόν. Η συζήτηση έληξε. Το Προεδρείο έχει λάβει μία πρόταση ψηφίσματος και η σχετική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30 ε, το πρωί. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες που συνιστούν διακρίσεις σε βάρος λιθουανικών φορτηγών στα ρωσικά σύνορα. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην ε, συντάκτη της προφορικής ερώτησης, τη συνάδελφο Γκέσιν Μέισνερ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όντω, είναι γεγονός. Αυτά που συμβαίνουν τώρα στα σύνορα Λιθουανίας-Ρωσίας ε, δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε καμία περίπτωση από πλευρά μα. Η Λιθουανία έχει 650 ε, εταιρείε μεταφορικέ με 13.000 ε, φορτηγά που μεταφέρουν πάρα πολλά εμπορεύματα στη Ρωσία. Και πρόσφατα η Ρωσία έχει σαγάγει ειδικού τελωνιακού ελέγχου για τα λιθουανικά φορτηγά. Αυτό είναι μέτρο αντιπίνων. Και για τα ΙΧ μάλιστα έκαναν ιδιαίτερου ελέγχου στους Λιθουανούς χωρίς καμία αιτιολόγηση. Καψώνει είναι ουσιαστικά και μάλιστα χρειάζονται και του ζητάνε και ειδική συνοδεία ε, τα φορτηγά αυτά στη ρωσική επικράτεια. Αυτό δεν μπορούμε να το ανεχθούμε με κανέναν τρόπο γιατί η Λιθουανία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα αυτό αφορά συνολικά το ίδιο μεταφορές στην Ένωση και στις γειτονικές χώρες. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι από το 2012 η Ρωσία είναι μέλος του ΠΟΕ, αντίστοιχα έχει δεχτεί τους όρους που ισχύουν και όλα αυτά δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με την κατάσταση. Βέβαια, οι λιθουανικές εταιρείες τώρα έχουν πολλές ζημίες, 2 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα περίπου από αυτές τις κατεστερήσεις και την παρελκυστική τακτική ε, και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι αυτό να παραμένουμε θεατές. Είναι σαφές ότι η Ρωσία προσπαθεί τώρα πρώην Σοβιετικές χώρες που είναι μέλη της Ένωσης ή κοντά στην Ένωση να τις τιμωρήσει με κυρώσεις. Το έχουμε ξαναδεί αυτό σε άλλα κράτη-μέλη ή άλλα υποψήφια, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία και εκεί ε, έχουν αντίστοιχη τακτική οι Ρώσοι. Μπορώ να σας διαβάσω αυτό που είπε ο πρόεδρος της ομάδας μας, ο Γκίφερ Χόφστατ, ε, με ε, τις διακρίσεις εις βάρος Λιθουανών οδηγών φορτηγών είτε διακρίσεις σε βάρος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνατε τίποτα, προτίθεστε να κάνετε κάτι για να αποτραπεί αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Μάισνερ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας από τον συνάδελφο Ιμπράσας. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Ναι, οι ιδέες που ε, συμμεριστήκατε μαζί μας ε, σύμφωνα με την ομάδα EFD η ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο αυστηρή στάση εφόσον η εξαγωγής της κρέατος της Λιθουανίας έχουν, είχαν απώλειες, ζημίες, που είναι ζημίες όλων των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει όλη η Ευρώπη να μιλήσει με μία φωνή για να προστατεύσει την Λιθουανία. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομη. Βεβαίως συμφωνώ ότι θα πρέπει ε, να είμαστε ομόφωνοι απέναντι σε αυτό. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Ντεχούχ, τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη. Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τις αρχές της Λιθουανίας ότι οι τελωνιακές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στα συνοριακά φυλάκια από τις 12 Σεπτεμβρίου αυτού του έτους και αυτά τα μέτρα διέκοψαν το εμπόριο ε, και δεν συνδέονται με στόχους ε, κινδύνου. Πρόκειται για διακρίσεις και παραβιάσεις των κανόνων του ΠΟΕ. Στις 18 Σεπτεμβρίου ε, με τον συνάδελφο Σεμέτα έστειλα μια επιστολή στον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας Αλεξέη Γκουντουγκιάγεφ και στον Ανδρέα Γιαννίνοφ επικεφαλής των Τελωνίων τονίσαμε ότι τα μέτρα τα οποία θεσπίστηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου είναι ε, πηγή ανησυχίας από οικονομικής και νομικής απόψεως. Ζητήσαμε διευκρινήσεις σχετικά με τα μέτρα αυτά, εξηγήσει για τα μέτρα και κάναμε έκκληση στις αρχές για να άρουν αυτούς τους περιορισμούς μέχρι σήμερα οι ρωσικές αρχές δεν έδωσαν ε, διευκρινήσεις ε, σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτούς τους τελωνιακούς ελέγχους. Τώρα ελέγχουμε την συμβατότητα αυτών των μέτρων με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και κυρίως με το άρθρο 11 ε, της Γενικής Συμφωνίας ΓΚΑΤΣ για το εμπόριο και τους δασμούς. Για να δούμε αν ε, δικαιολογείται ο έλεγχος. Θα είναι επίσης σημαντικό να έχουμε πληροφορίες από τις λιθουανικές αρχές σχετικά με την αιτιολόγηση των μέτρων αυτών. Εν τω μεταξύ το θέμα αυτό θα μπει στην ατζέντα, στην ημερήσια διάταξη ε, του επόμενου Συμβουλίου ΠΟΕ που θα λάβει χώρα στις 18 Οκτωβρίου στη Γενέβη ως δυνητική παραβίαση των κανόνων του ΠΟ. Επίσης θα συζητηθεί πριν σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Ρώσους ομολόγους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο θα ήταν να εξετάσουμε την, το πολιτικό σκέλος αυτού του μέτρου σε σχέση με, τις, με τους πρόσφατους περιορισμούς στα γαλακτοκομικά προϊόντα της Λιθουανίας δεν ενημερωθήκαμε ε, σχετικά με αυτά τα προϊόντα από τη Ρωσία. Η Επιτροπή έχει εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των λιθουανικών γαλακτοκομικών υπάρχει, που παρέχουν μεγάλη προστασία καταναλωτών. Αυτό το πλαίσιο διατροφικής ασφάλειας εξασφαλίζεται με επιθεωρήσεις της Επιτροπής και με ένα σύστημα έγκαιρου προειδοποίησης ε, για δράση σε περίπτωση που ένα προϊόν θεωρηθεί μη ασφαλές. Υπάρχουν διαφορές ε, ανάμεσα στα πρότυπα της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε μερικές περιπτώσεις πιστεύουν ότι τα πρότυπα δεν είναι αναγκαία για την προστασία των καταναλωτών. Γι' αυτό η Επιτροπή έκανε έκκληση στις ρωσικές αρχές για ανάλογη δράση ε, ε, σχετικά, ε, σε σχέση με τα δικά της προϊόντα και τα προϊόντα της Λιθουανίας. Οποιοδήποτε περιορισμός που βασίζεται σε υγειονομικούς λόγους θα πρέπει να δικαιολογείται και να λεχθεί ποιο είναι η απειλή και οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες με τον κίνδυνο. έχουμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο αύξηση των κυρώσεων. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τους εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη δέσμευση προς τον ΠΟΕ. Με βάση περαιτέρω πληροφορίες και εξελίξεις θα συστήσω στο σώμα ε, μέτρα σύμφωνα με την, τη Γενική Συμφωνία του ΠΟΕ για το εμπόριο και τους δασμούς. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και θα δώσω τον λόγο στον συνάδελφο Κάσπαρη του ΕΛΚ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε, αλλά ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά με τρόπο πολύ τεχνικό και πάρα πολύ εύκολο, γιατί τη ζούμε εδώ και μερικές εβδομάδες. Από ό,τι φαίνεται η Ρωσία ποντάρει όσο μπορεί να τορπιλήσει την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Αυτό είναι ένα και μόνο παράδειγμα που μα απασχολεί σήμερα. Ξαφνικά μεταφορικέ εταιρείε με φορτηγά από τη Λιθουανία υφίστανται αυτή τη μεταχείριση στοχευμένα. Το δεύτερο είναι πολύ πρόσφατο. Χθε το πρωί τα γαλακτοκομικά που δεν θέλουν. Καλό είναι να το φέρετε στον ΠΟΕ, αλλά επιγόντως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβληματιστεί μήπω να καλέσει ε, τον ε, Ρώσο πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συνομιλίες και θα χαιρόμουν και με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και τους άλλους που έχουμε ε, στη Ρωσία να πούμε ξεκάθαρα στους Ρώσους ότι οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας απειλούνται μαζικά και έχει και πολιτική διάσταση αυτό για τη συνεργασία μας και είναι άκρο επιζήμιο. Επίσης θα επιθυμούσα εδώ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να φύγει ένα σαφέ μήνυμα δεν ε, υφίσταται επίθεση η Λιθουανία, αλλά όταν με εμπορικά μέτρα κάποιο επιτίθεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα, επιτίθεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ επιθυμώ μια ευρεία ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Είναι από τα μικρότερα κράτη-μέλη μα και δεν θα πρέπει να εμοραγεί κυριολεκτικά. Υπάρχει προσεχώς μια μεγάλη σύνοδος κορυφής στη Λιθουανία με μεγάλα πολιτικά μηνύματα και δεν μπορεί ε, Ρωσία που είναι και τέρο μας ε, να έχει όμοιρο μια χώρα. Ε, θα πρέπει να έχουμε σαφή μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σαφείς δηλώσεις επιθυμώ από την ύπατη εκπρόσωπο. Να διατρανώσουμε στους Ρώσους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι Αφενός είμαστε υπέρ των καλών σχέσεων με τη Ρωσία και φίλοι του, αλλά από την άλλη να πούμε ξεκάθαρα ότι όποιος επιτίθεται σε μία χώρα τα βάζει με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε αλληλέγγυοι. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Κασπάρη. Και υπάρχει μπλε κάρτα από το συνάδελφο Μάισνερ. Συμφωνείτε, δέχεστε. Τι συνάδελφο Μάισνερ. Θα είμαι και πολύ σύντομη και γρήγορα. Αυτό με τα γαλακτοκομικά το είπατε και έχετε δίκιο. Και για τη Λιθουανία. Για τη Ρωσία δεν χάλασε ο κόσμος. Μπορούν να αγοράσουν γάλα και παλού. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, οι ε, εξαγωγέ της Λιθουανίας σε γαλακτοκομικά πηγαίνουν κυρίως στη Ρωσία. Αυτό δεν θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ακριβώ αυτό που λέτε είναι ε, τρομακτικό. Από ότι μια ε, επιβαρύνεται και ε, παθαίνει τεράστια ζημιά ο κλάδος των μεταφορών στη Λιθουανία, αλλά εξ όσων γνωρίζω το 90% των εξαγωγών γάλακτος ε, πηγαίνει στη Ρωσία. Δεν ξέρω καμία άλλη χώρα που να έχει προβλήματα με το λουθουανικό γάλα. Δεν το έχουν δηλώσει στο σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση στο ΡΑΠΕΞ. Ξαφνικά η Ρωσία ανακάλυψε ότι έχει πρόβλημα το γάλα τη Λιθουανία. Ευχαριστώ. Το πολύ η συνάδελφο Μπλίνκεβιτσούτε από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ε, Κύριε Επίτροπε, Είμαι ευγνώμων για την ε, θέση της ε, Κομισιόν στα, πέραντι στα μέτρα ε, διάκρισης που εφαρμόζει η Ρωσία εδώ και αρκετό καιρό. Σας καλώ να λάβετε άμεσα όλες τα απαραίτητα μέτρα και να προβείτε τις απαραίτητες ενέργειες γιατί ακόμα δεν ε, ήταν αποτελεσματικά. Ε, λόγω της κατάστασης στα σύνορα έχουμε τεράστιες απώλειες. Η κατάσταση με τα γαλακτοκομικά ζημιώνει ε, τους παραγωγούς μας ε, και με τη σειρά του αυτό θα επιβλάψει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όλα αυτά γίνονται κατά τη διάρκεια της, ε, της Προεδρίας της Λιθουανίας όταν ταυτόχρονα προετοιμάζουμε τη διάσκεψη κορυφής στο Βίλνιους. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ενωμένη πολιτική απάντηση στις ενέργειες αυτές κατά της Λιθουανίας. Σας θαρρύνω λοιπόν να σταματήσετε, να θέσετε ένα τέλος σε αυτές τις ε, ε, διαδικασίες. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται τέτοια μέτρα κατά άλλων χωρών, στο, άλλων χωρών στο μέλλον. Και κυρία Πρόεδρε, τώρα θα ήθελα να κάνω έκκληση προς εσάς. Ε, ο Αντιπρόεδρος της Λιθουανίας, ο κύριος Λεσκάλετσε, συμμετέχει στη συνεδρίασή μας. Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε τη γνώμη του. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα λεπτό για εκείνον, για να μπορέσει και εκείνος να πάρει το λόγο. Πρόεδρος. Εάν ο αντιπρόεδρο της κυβέρνηση επιθυμεί να πάρει το λόγο, βεβαίω, ε, και είναι πρόσδεκτος. Θέλετε να σχολιάσετε, θέλετε να παρέμβετε. Yes, Okay. Ναι, το επιθυμώ. Μπορώ τώρα αμέσω να πάρω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Αντίθετα από ότι ήθιστε σε αυτή την αίθουσα, μιλώ ως εκπρόσωπος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και όχι ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου, αλλά εκ μέρους της χώρας μου. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία, σας ευχαριστώ Επίτροπε, σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό. Σας ευχαριστώ που κάνετε αυτή τη συζήτηση και ελπίζω πως ε, θα προβείτε σε ενέργειες και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες πτυχές που ε, δημιουργούν ανησυχία όχι μόνο στη Λιθουανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί πρόκληση για όλους μας. Είναι πρόκληση για το σύνολο του εμπορικού ε, συστήματος και τους κανόνες του ΠΟΕ. Όπω γνωρίζετε η Ρωσική Ομοσπονδία χωρί καμία προηγούμενη ειδοποίηση όπως θα έπρεπε, χωρί καμία εξήγηση επίση, εφαρμόζει περιορισμούς εδώ και αρκετό ε, καιρό. Περιορισμούς ε, στους λιθονούς μεταφορείς και όχι μόνο στους λιθονούς αλλά και στα αγαθά που μεταφέρουν οι λιθουανοί μεταφορείς προς την Ρωσική Ομοσπονδία και απλώ φορτώνονται στη Λιθουανία, δεν παράγονται στη Λιθουανία. χωρί κανένα λόγο όπως σας είπα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Είναι κάτι που δεν είναι φυσιολογικό και είναι ενάντια σε οποιοδήποτε κανόνα. Σε οποιαδήποτε αρχή φυσιολογικής συνύπαρξης. Η Ρωσία δεν περιορίζεται όμως αυτό. Άρχισε να εισάγει και απαγορεύσεις. Ξεκίνησε δηλαδή μια δημόσια εκστρατεία κατά της Λιθουανίας και της γαλακτοκομικής της παραγωγής και κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει, τι θα γίνει εάν δεν αντιδράσουμε. Μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή. Πρόκειται για μια πρόκληση όχι μόνο για την Λιθουανία, αλλά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και εκτιμάμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες και τις αντιδράσεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Σε αυτή τη χρονική φάση η αλληλεγγύη με την Λιθουανία είναι η μίνιμουμ στήριξη που μπορεί να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη οφείλει να το κάνει αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την αντίδρασή σας και σας ευχαριστώ για την αλληλεγγύη σας. Η σας ευχαριστώ κύριε Λεσκεβίσιους που είστε Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μιλήσατε εξ ονόματος της ε, Λιθουανίας. Ε, και τώρα δίνω το λόγο στον συνάδελφο Ζήλε, εξ ονόματος της ΕΣΥΑΡ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ε, διατέλεσα υπουργός και ε, επιβλήθηκε εμπάργο στις λετονικές εξαγωγές προς την ε, Ρωσία. Ε, και ξέρουμε ότι και στην Εστονία υπήρξαν προβλήματα σε σχέση με ένα μνημείο κτλ. Τώρα ήρθε η σειρά της Λιθουανίας. Ε, και στην ενέργεια και στις μεταφορές υφίστανται διακρίσεις σε ευρωπαϊκές χώρες από τη Ρωσία. Αυτά τα γνωρίζουν όλοι οι παρόντες και για ποιο λόγο δρά ε, με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία και στρέφεται κατά της Λιθουανίας. Διότι ως πρώην Σοβιετική Ένωση θεωρεί τις χώρες αυτές ε, δικά της χωράφια και ε, έχει οθετήσει και την αρχή διέρη και βασίλευε και θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κάτσει τώρα να υπερασπιστεί μία χώρα. Μια χώρα όμως σαν τη Λιθουανία αυτή τη στιγμή είναι και ε, στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα πει η Φίλιος αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύσει τη χώρα της Προεδρίας. Ευχαριστώ. Δέχεστε από τον κύριο Λάιχτφριντ μια ερώτηση, γαλάζια κάρτα. Παρακαλώ, ο κύριος Λάιχφριντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζήλε, έχω την εξή ερώτηση. Ο πολιτικός σα σχηματισμός συνήθως είναι αρκετά επικριτικός ε, όταν η Ευρώπη έχει ενιαία θέση. Και γενικά δεν είστε πάρα πολύ υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εδώ δεν είναι ευκαιρία να φανεί ότι μια ενωμένη Ευρώπη μπορεί να είναι πιο ισχυρή προς τα έξω από μια κατακαιρματισμένη. Μπορείτε να τα πείτε λίγο αυτά και στους συναδέλφους πολιτικής ομάδας και να τους πιέσετε. Ευχαριστώ κύριε Θέλω να πω ότι η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών είναι πάρα πολύ υπέρ ε, μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Ε, είμαστε υπέρ αυτών των αρχών και ξέρουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά. Αυτό είναι ένα θέμα διακρίσεων κατά της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό δεν είναι αντίφαση με τις δικές μας θέσεις. Ανέκαθεν ήμασταν υπέρ της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, εμείς είμαστε κατά της Ομοσπονδιακής Φεντεραλιστικής Ευρώπης. Θα θέλω να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Αντρίκενε για δύο λεπτά. Ναι, συζητούμε εδώ αυτές τις κατάφορες παραβιάσεις της Ρωσίας που δεν είναι αιτιολογημένες και είναι κατά της Λιθουανίας που είναι μέλος της εσωτερικής αγοράς. Η Λιθουανία έγινε μέλος του η Ρωσία έγινε μέλος του ΠΟΕ πέρσι, παρόλα αυτά δεν τηρεί τις δεσμεύσεις από τις 11 Σεπτεμβρίου. Η Ρωσία έχει επιβάλει μέτρα διακρίσεων κατά της Λιθουανίας και τα αιτήματα της κυβέρνησης της Λιθουανίας παραμένουν χωρίς απάντηση. Έχουμε αλαζονικές ε, ε, δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης από την Ρωσία. Θα πρέπει η Ρωσία να λογικευθεί έχουμε λάβει απειλές ότι η Ρωσία θα επιβάλλει εμπάργο πάνω στα γαλακτοκομικά προϊόντα και ότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί ενδελεχείς έλεγχοι στα προϊόντα, τα αλλιευτικά και στα κρέατα. Η Ρωσία ε, δεν προσπαθεί να χαλαρώσει την πίεση. Πρέπει η αντίδρασή μας να είναι αυστηρή θα πρέπει η Ρωσία να παράσχει δικαιολογία, εξηγήσει σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί έλαβε αυτά τα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να απευθυνθεί στον ΠΟΕ ούτως ώστε ο ΠΟΕ να ζητήσει από την Ρωσία να ε, τηρήσει τους κανόνες του ΠΟΕ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ε, υπάρχουν ασύμετρα μέτρα. Το θέμα Μακνίτσκι. Σήμερα είναι η Λιθουανία, αύριο μπορεί να είναι ένα άλλο κράτος μέλος που θα πληγεί. Δεν μπορούμε αυτό να το ανεχθούμε. Επίτροπε, συνάδελφοι, πριν από δύο εβδομάδε μιλήσαμε για τα ε, διακριτικά μέτρα τη ρωσική ομοσπονδία απέναντι στου ανατολικού μα ε, ε, γείτονε. Σήμερα συζητάμε τα διακριτικά μέτρα τη ρωσική ομοσπονδία έναντι των δικών μας κρατών μελών, του κράτου μέλου μάλιστα που έχει την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Λιθουανία. Και πιστεύω πω αυτό είναι απαράδεκτο. Η ρωσική συμπεριφορά είναι για μας, για του σοσιαλδημοκράτε, απαράδεκτη. Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο, δεν θέλουμε να ορθώσουμε νέους φραγμούς, αντίθετα θέλουμε συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ναι, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό οικονομικό χώρο όπου η Ρωσία είναι στρατηγικός μας εταίρος. Αλλά, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να περιμένουμε και να δεχτούμε μάλλον τέτοιου είδους συμπεριφορά. Οπότε στηρίζουμε απόλυτα τους Λιθανούς συναδέλφους και εκφράζουμε την πλήρη μας αλληλεγγύη με τη Λιθουανία. Συμφωνώ απολύτως ότι δεν είναι μόνο μια επίθεση προς τη Λιθουανία, είναι μια εμπορική επίθεση εναντί ολόκληρης της Ένωσης και θα ήθελα να ζητήσω και εγώ από τον Επίτροπο να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του εντός του ΠΟΕ και εκτός του ΠΟΕ ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είναι απαραίτητο μάλιστα να γίνει αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί οι παραγωγοί, οι αγρότε, στη Λιθουανία πλήττονται πολύ σοβαρά και δεν μπορούμε να ανοιχτούμε τέτοιου είδου συμπεριφορά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρούσικ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να νιώθουμε όλοι ικανοποίηση που η Ευρωπαϊκή μας Ένωση γίνεται ουσιαστική και πιο εδρεωμένη ένωση. Και συνεχίζεται αυτό και χάρη στην ενοποιημένη ενεργειακή πολιτική και την κοινή πολιτική γειτονίας προς την Ανατολή. Ε, υποτίθεται ότι οι γείτονες είναι φιλικοί και συνεργάσιμοι. Αλλά όχι μόνο αυτό δεν είναι, αλλά είναι και εχθρική. Αυτή είναι η σημερινή Ρωσία. Απέναντι στις πρώην υπηρετικές της ε, ε, απικίες που βλέπει να στρέφονται όλο και πιο ε, πολύ προς την Ευρώπη και όχι την Ασία ή την Ευρασία. Έχει θυμώσει που οι έκπτωτες Μητροπόλεις της τώρα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου η Λιθουανία προσπαθούν να καταστρέψουν την οικονομία μας με τις επικοινωνίες, με τις μεταφορές και είναι πρόκληση για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή συζήτηση θα πρέπει να αφορά περισσότερο όχι τα λιθουανικά φορτηγά στα ρωσικά σύνορα, αλλά την ανώμαλη κατάσταση στα σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Δεν είναι εμπορικές σχέσεις Ρωσίας-Λιθουανίας, αλλά Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας εμπορικές σχέσεις. Και ταυτόχρονα οι απώλειες και οι ζημίες είναι ευρωπαϊκές, όχι λιθουανικές. Οι λιθουανικές εταιρείες είναι ευρωπαϊκές. πραγματική πολιτική θα σήμαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιραστεί και επιμεριστεί τις ζημίες ε, που υφίσταται η Λιθουανία λόγω των ανατολικών πολιτικών. Ο συνήθως θεωρεί το Κρεμλίνο ότι μπορεί να επιτίθεται στα κράτη-μέλη της Ένωσης αγνώντας την ίδια την ύπαρξή της. Λάθος εικόνα δίνουν δίνουμε εμείς. Είναι διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα δεν είναι όσο ενωμένη θα έπρεπε. Θα πρέπει να παρέλθουν αυτοί οι καιροί και να έρθει ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαντσπέργης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω από την κρίση χρέους και την οικονομική θα πρέπει να ισχύει εξής αρχή παγκοσμίως. Όποιος επιτίθεται σε μια χώρα της Ευρώπης, επιτίθεται στην Ευρώπη ολόκληρη. Είτε είναι αυτή η Ελλάδα που επιτέθηκαν οι κερδοσκόποι σε αυτήν. Είτε πρόκειται για τη Λιθουανία που της επιτέθηκε μια πρώην υπερδύναμη. Νομίζω τα ίδια θα πρέπει να ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, όπως και με την οικονομική κρίση και τη χρηματοπιστωτική. Δεν είμαι όμως βέβαιος εάν μπορούμε με εμπορικά μέτρα ή αποκλειστικά εμπορικά μέτρα να αντικρούσουμε κάποιες τέτοιες επιθέσεις που έχουν να κάνουν με εξουσίες και δυνάμεις. Όταν αρχίζουν τέτοια παιχνιδάκια, είτε η Ρωσία είτε όποιος άλλος, να παίξουμε κι εμείς, να δουν κι αυτοί πώς το παίζουμε το παιχνίδι και να είμαστε πιο δραστήριοι και πιο ενεργοί στην ε, αντεπίθεση. Επίτροπε, έχετε μια πολύ ωραία φήμη τώρα στην Κίνα. Μήπως να έχετε και την ίδια στη Ρωσία προσεχώς. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, colleague Περνάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διαδικασία Catch the Eye. Και πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μόρκενάιτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τις ανησυχίες ε, για την Λιθουανία. Δεν είναι μόνο θέμα της ε, Λιθουανίας. Η Ρωσία έχει ήδη απαγορεύσει τα γαλακτοκομικά προϊόντα και απείλησε να κάνει το ίδιο με τα αλλιευτικά προϊόντα και τα κρέατα. Δεν, δεν καταλαβαίνουμε το πλαίσιο όταν βλέπουμε άλλους γείτονες που υφίστανται τις ίδιες πιέσεις, αλλά η Λιθουανία έχει τώρα διαπραγματεύσεις με την Κάσπρομ. Για, για θυμηθείτε τον ε, αγωγό Ντρούστα, ε, το πρόβλημα για την Λιθουανία Αυτές τα μέτρα είναι παραβίαση της αρχής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αναλογικότητας. Η Ρωσία είναι μέλος του ΠΟΕ. Η Ρωσική Ομοσπανδία θέλει νέες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή η συμπεριφορά μας κάνει να αμφιβάλλουμε αν μπορεί να ακολουθήσει τις δεσμεύσεις. Αύριο Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με τη Λιθουανία. Χρειάζεται η αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Κύριε Επίτροπε, εσείς επίσης είπατε ότι για κάποιο λόγο η Ρωσία εισήγε στάνταρ τα οποία επιστημονικώς δεν στέκουν. Ε, αυτό σημαίνει πως η Ρωσία είχε εδώ και καιρό σχέδια για να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στις χώρες μας ή σε οποιαδήποτε χώρα. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι πριν από τα Χριστούγεννα η Λιθουανία και η, Βαλ... η οι μεταφορείς της Βαλτικής ε, είχαν ε, δυνατότητα περάσματος ε, να διανύσουν μάλλον τη ρωσικά σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε την πολιτική οικονομικής προστασίας των στρατηγικών συμφερόντων των χωρών μας. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά που συμβαίνουν τώρα είναι αντίπεινα της Ρωσίας. Η Ρωσία ε, τιμωρεί τη Λιθουανία λόγω της πολιτικής ανατολικής γειτονίας και προσπαθεί να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει προσπαθώντας να πιέσει την γειτονική της χώρα. Μετά από την οικονομική μπλοκάζ που υπέστη η Λιθουανία το δεκαετία του 90, τώρα είναι η δεύτερη φορά που παθαίνει το ίδιο, μόνο που τώρα είναι χώρα της Ένωσης και τώρα πρέπει να κάνουμε έκκληση στην παλιά Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τίποτα δεν μπορεί να σταθεί μόνο του. Είναι επίθεση εναντίον της Ένωσης και γι' αυτό εκτιμώ την αλληλεγγύη των συναδέλφων και την, ε, τις παρατηρήσεις τους που είπαν ότι ε, πρέπει να αντιδράσουμε σαν να δεχόταν επίθεση η Ένωση ή να δεχόταν εκβιασμό ή άλλες επιθετικές δράσεις. Γι' αυτό πριν από τη διάσκεψη κορυφή του Βίλνιου και πριν να γίνουν σημαντικές δράσεις στην Ένωση θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην ξανασυμβεί. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κέλαμ. Ευχαριστώ. Είναι απαράδεκτη η πίεση αυτή, όχι μόνο εναντίον ενός κράτους μέλους, αλλά εναντίον όλων των χωρών. Και θα πρέπει ε, να θεωρηθεί ως εχθρική ε, στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι το διμερές και αυτό δεν συνέβη τυχαία παρόμοιες ε, βίες οικονομικές πιέσεις εφαρμόστηκαν για την Μολδόβα και την Ουκρανία. Θα πρέπει να λαμβάνουμε κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε ότι τα μέτρα της Ρωσίας είναι κατάφορη πολιτική πίεση. Χρειαζόμαστε ειδικά μέτρα από την Επιτροπή. Η πολιτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ρωσίας δεν είναι ε, φιλική και εμπνέεται από μετα-ιμπεριαλιστικές αρχές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σήμα αλληλεγγύης ότι είμαστε ενωμένοι για να υπερασπιστούμε τα κράτη-μέλη και να υπερασπιστούμε την ελευθερία των κρατών αυτών που θέλουν να ενταχθούν στη δημοκρατική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής γεγονός. Μιλούμε για διακρίσεις στη Ρωσία απέναντι σε μεταφορικές εταιρείες από τη Λιθουανία. Μεν, πλην όμως αυτές οι πρακτικές στη Ρωσία επαναλαμβάνονται. Και αυτό δεν στρέφεται μόνο κατά των χωρών της Βαλτικής. Υπάρχουν αντίστοιχες ε, ε, ρυθμίσεις και περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν σε κατασκευαστές και ε, ιδιοκτήτες ε, φορτηγών και μεταφορικές εταιρείες από την Πολωνία και αφορούσαν γαλακτοκομικά, ε, κρέας ή τυρί, γάλα και σε κάθε τέτοια περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει τη χώρα που υφίσταται τις διακριτικές πρακτικές και θα πρέπει να μιλήσουμε μία φωνή, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν χώρε που είναι περισσότερο λιγότερο σπουδέ. Και τέλο ο συνάδελφο Πάσκα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Η μη προαναγγελθήσα ε, μη μάλλον προαναγγελθείς έλεγχος, αυστηρότερος έλεγχος των εισαγωγών είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για πολλές χώρες. Τα εμπορεύματα που μεταφέρει, μεταφέρουν οι μεταφερείς της Λιθουανίας προέρχονται από άλλες χώρες της Ένωσης και γι' αυτό οι περιορισμοί αυτοί ε, πλήττουν και τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Η Ρωσία είναι βασικός ε, ε, εμπορικός εταίρος και άρα ε, θα έπρεπε κανονικά τα μέτρα αυτά να είναι προς το κοινό συμφέρον. Ε, δεν υπάρχει η λύση δεν έγκυται σε μονομερείς αυτές τις δράσεις από πλευράς της ρωσικής πλευράς. Θα πρέπει λοιπόν μέσω της διπλωματίας μας να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα κλιμακωθούν όλα αυτά σε βασικά οικονομικά προβλήματα με σημαντικές επιπτώσεις για τις οικονομίες μας. Είμαι πεπισμένος επίτροπε ότι δεν θα πρέπει να διστάσουμε και να αρχίσουμε να μιλάμε ουσιαστικά με τους Ρώσους ομολόγους μας. Ευχαριστούμε κύριε Πάσχη και τώρα Επίτροπε Ντεγκούχτε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, υπάρχουν μερικές αμφιβολίες στο μυαλό μου ότι τα μέτρα αυτά έχουν πολιτικά κίνητρα και μάλλον ε, συνδέονται με τις ανησυχίες ε, της Ρωσίας σχετικά με την πολιτική της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Παρακολουθώντας την συζήτηση, νομίζω ότι αυτό σκέφτεστε κι εσείς, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν είναι επειδή υπάρχουν πολιτικά κίνητρα που δεν θα πρέπει να προετοιμαστούμε δεόντως πρωτού πάμε στον ΠΟΕ. Και αναλύουμε τώρα την συμβατότητα με τον ΠΟΕ αυτών των μέτρων. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να πάμε στον ΠΟΕ αν δεν έχουμε μια καλή ανάλυση που να βασίζεται σε γεγονότα και στατιστικές. Στις 18 Οκτωβρίου έχουμε το Συμβούλιο του ΠΟΕ για τα αγαθά και θα αναφέρουμε το θέμα αυτό. Και το στις 18 θα έχουμε συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο και πριν από τις 18. εγώ είμαι νομικός και Προτού πάει κανείς σε ένα δικαστήριο, το, το ΠΟΕ είναι, ο ΠΟΕ είναι δικαστήριο, ετοιμάζει κανείς την όλη δικογραφία, το φάκελο της περίπτωσης, όλες οι περιπτώσεις που υποβάλλονται στον ΠΟΕ είναι αιτιολογημένες, τεκμηριωμένες αυτές οι υποθέσεις και γι' αυτό δεν χάνουμε καμιά υπόθεση γιατί θα κάνουμε και το ίδιο και βασιζόμαστε στην συνεργασία της Λιθουανίας για το σκοπό αυτό. Μπορεί κανείς να αντιδράσει πολιτικά σε τέτοια μέτρα. Και ο κύριος Κασπάρη ανέφερε τη δυνατότητα να καλέσουμε τον Ρώσο πρέσβη. Θα μπορούσα να το κάνω τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει πρόβλημα και νομίζω ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές τους Ρώσους, όπως είπατε πολύ, ότι όταν κανείς ε, λαμβάνει τέτοια μέτρα εναντίον ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαν λαμβάνει μέτρα εναντίον όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν έχω καμία μαγική λύση για να επιλύσω το πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη. Έχω έναν κατάλογο όλων των προβλημάτων που είχαμε με τη Ρωσία από τις 20 Μαρτίου 2012 όταν υπήρξε απαγόρευση ε, για κτηνοτροφικά ε, προϊόντα από όλες ε, τις ευρωπαϊκές λόγω του ιού Σμόλεμπεκ. Από τότε υπάρχει ένας κατάλογος 10 μέτρων που έλαβαν ε, οι Ρώσοι εναντίον πολλών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο εναντίον των Λιθουανών. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το νέο και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, αλλά θα ήθελα να κατανοήσετε ότι αυτό πρέπει να γίνει με βασικές αποδείξεις που θα πρέπει να συλλέξουμε και θα θα, ήθελαμε να, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τους Ρώσους γιατί το κάνουν αυτό, πώς και γιατί και με βάση όλο το υλικό που θα έχουμε θα λάβουμε σύντομα τις δέουσες αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Και συνεχίζουμε με την έκθεση του Malcolm Harbour Σκάφη «Αναψυχής και ατομικά».